Λοιπόν, επαναλαμβάνει η συνεδρίαση, η διακοπήσα. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης είναι στη διάθεσή σας. Έχετε παρατηρήσει όσον αφορά τη χθεσινή συνεδρίαση και τα πρακτικά της. Όχι, γιατί αυτή η περιπτώση θεωρούνται συγκεκριμένα τα πρακτικά.